για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τη δική μας συνεδρίαση, γιατί έχω και πολλές ε, ανακοινώσεις που θα μας... Ε, το παλιό, το παλιό. Φάνε αρκετό χρόνο. Και 10 και 4 πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Καταρχήν για την ημερήσια διάταξη. Στο σημείο 5, στην ενημέρωση για τις διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις, θα σας ενημερώσω για τον τριμερή διάλογο για τους έμμονους ή επίμονους οργανικούς ρήμπους που έγινε την Τρίτη. Με αυτή την αλλαγή λοιπόν μπορούμε να εγκρίνουμε την ημέρη σε διάταξη, όχι από ό,τι φαίνεται, οπότε εγκρίνεται. Στα έγγραφα της συνεδρίας θα βρείτε και την έκθεση της αποστολής αντιπροσωπής ΕΜΒΗ στην διάσκεψη κορυφής που έγινε 12 με 14 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο ε, με πρωτοβουλία του Τζέρι Μπράουν, του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, προκειμένου να ενισχυθούν οι παγκόσμιες δεσμεύσεις υπέρ του κλίματος εν ώψη της COP28 στο, στο Κατοβίτσε. Επίσης ακυρώνεται η συνεδρίαση πρωί και απόγευμα και η έκτακτη συνεδρίαση για τα δάση, Άγκρη και Έμβη, παρουσία του Επιτρόπου Χόγκαν, θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο, 7 το απόγευμα. Σήμερα έχουμε 20 γλώσσες διερμηνία και φυσικά ως συνήθως έχουμε μοιράσει ε, ηλεκτρονικά τα θέματα της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου πριν και απόγευμα, όπως σας είπα, ακυρώνεται και έχουμε και μετάδοση στο διαδίκτυο. Πρακτικά, πρακτικά τη 25 η Οκτωβρίου 2018, αν μέχρι το τέλος συνεδρίε δεν υποβληθούν παρατηρήσει, θα θεωρηθούν συγκεκριμένα τα πρακτικά. Ενημέρωση τώρα για τις τρέχουσες διοργανικέ διαπραγματεύσεις. Τέσσερι πληροφορίε θα σας δώσω. Καταρχήν, για την επισήμανση των ενοπνευματοδόμποτων. Τρίτο άτυπο τριμερή διάλογο έλαβε χώρα στι 27 Νοεμβρίου και μετά από πολλή προσπάθεια μπορώ να σας ενημερώσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι καταλήξαμε σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για όλα τα πολιτικά θέματα στην πρόταση αυτή για την επισήμαση των αλκοολούχων των νοπνευματοδών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα τρία εκκρεμή πακέτα και έχουμε μια προκαταρκτική συμφωνία που θα ε, ψηφιστεί στις 22 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας. Και στις 10 Δεκεμβρίου στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας. Εν τω μεταξύ, οι θα κοινοποιηθούν από την Επιτροπή στην ε, Ειδική Επιτροπή Τεχνικών Φραγμών για το εμπόριο του ΠΟΕ και θα έχουν δύο μήνες για την εξέταση περάμε τώρα στο θέμα των πλαστικών. Είχαμε το δεύτερο τριμερή διάλογο στις 28 Νοεμβρίου. Μια προσωρινή συμφωνία επετεύχθη για πολλά θέματα, για τα άρθρα 1 και 10, καθώς και για πολλούς ορισμούς. Η Προεδρία επισήμανε την σύγκληση προς το Κοινοβούλιο για τα, για τα λευτικά εργαλεία, το περιεχόμενο των μπουκαλιών ποτών, τα προϊόντα πολυστηρένης, τα φίλτρα του καπνού και για να διευκολύνουμε τη συζήτηση υποβάλαμε συμβαστικές τροπολογίες για πέντε άρθρα καθώς και τους περιορισμούς της αγοράς και, μείωση, και μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης μεταξύ άλλων. Σημειώθηκε πρόοδος για το άρθρο 5 που αφορά τους περιορισμούς στην αγορά και το παράρτημα Β όπου Συμβούλιο και Κοινοβούλιο συμφώνησαν να διευρύνουν την κατηγορία των προϊόντων για τα, ε, με πολυστηρένα να, να απαγορευτούν και συμφώνησε να εξετάσει περαιτέρω πιθανές συμβαστικές τροπολογίες και να συμπεριλάβει τα οξιαπικοδομήσιμα προϊόντα στο κατάλογο των απαγορευμένων προϊόντων, δεχόμενο τις ε, εξαιρέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσθέτοντα απαγόρευση για τα 100% πλαστικά κύπελα προκειμένου να διαφυλάξει τη φιλοδοξία του κειμένου. Σε ό,τι αφορά τα ε, οχήματα και φορτηγά με εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είχαμε τον τρίτο τριμέρι διάλογο στις 4 Δεκεμβρίου, πριν από λίγες μέρες την Τρίτη, και Προσωρινά έχουμε κλείσει κάποια θέματα όπως τα, τις μετρήσεις WLTP, την σήμαση για φορτηγά και αυτοκίνητα, ε, το κανονισ... τους στόχους του κανονισμού άρθρο 1, ε, το πεδίο εφαρμογή, τα οχήματα νη 1, το άρθρο 2, τις ειδικέ εξαιρέσει, ε, την παράταση μέχρι το 2028 και κάποιες αιτιολογικές σκέψεις υπέρ του περιβάλλοντος έγιναν ανταλλαγές απόψεων, για τους μετρητές κατανάλωση καυσίμων και τη δίκαιη μετάβαση, την ενδοϊπηρεσιακή συμμόρφωση, το, την ανάλυση του κύκλου ζωής και την οικολογική καινοτομία. Παρ' όλα αυτά δεν κατα, καταλήξαμε σε συμφωνία, απλώς έγινε συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τα βασικά θέματα των στόχων και των οχημάτων μηδενικών εκπομπών και τα σχετικά ενάψματα, οι δύο συνομοθέτες Δυστυχώ έχω μεγάλη απόκληση και διαφορά στι απόψει του και μια και δεν έγινε καμία κίνηση από το Συμβούλιο, περιμένουμε την ε, συνάντηση τη παρασκευή και προτείνουμε νέο τριμερή διάλογο τη Δευτέρα στο Στρασβούργο που κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει στι 9 το βράδυ. Τελευταίο θέμα ε, για το οποίο θα ήθελα να σα ενημερώσω είναι αναδιατύπωση για του έμονου η επίμονου Οργανικού ρήπου. Ο πρώτο άτυπο τριμερής διάλογο έγινε επίση 4 Δεκεμβρίου. Εξετάστηκε το σύνολο του κειμένου με ε, καταρχήν συμφωνία για πολλά πολιτικά θέματα, όπως ε, τα νέα καθήκοντα του Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Βέβαια, το βασικό θέμα που αφορά τα μέσα για την τροποποίηση των παραρτημάτων όπου το Συμβούλιο πρότεινε αντικατάσταση των κατεξουδότηση πράξεων με την τακτική νομοθετική διαδικασία σε ό,τι αφορά τα παραρτήματα 1 και 2 και διαγραφή των ορίων συγκέντρωσης που αναφέρονται στα παραρτήματα 4 και 5 με την έγκριση των τιμών αυτών με εκτελεστικές πράξεις αυτό δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνο. Η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου εξέφρασε τις ανησυχίες και τη δυσαρέσκειά του με την προσέγγιση του Συμβουλίου για πολιτικού θεσμικού και νομικού λόγου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση εξέφρασε ανησυχίε και γενικώ στήριξε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Εν ώψη λοιπόν όλων αυτών, ε, η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε την ε, προθυμία να συμμετάσχει σε δεύτερο και ενδεχομένω τελικό οριστικό τεμερι διάλογο 18 Δεκεμβρίου, υπό τον όρο όμω ότι το Συμβούλιο θα δείξει προθυμία και ελαστικότητα να αναθεωρήσει είναι εντολή του στα θέματα αυτά. Τέλος, για διάφορα θέματα έγινε παραπομπή σε τεχνικό επίπεδο συζητήσεων. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις και περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. So I hope you prepared your voting. Ελπίζω να έχετε ετοιμάσει τις ε, κάρτες ψηφοφορίας ε, και τώρα θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία για την γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση εφαρμογής, ε, σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά τους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κύριε Γιάβορ, θα θέλατε μήπως να ανεβείτε εδώ. Επειδή με μπερδεύετε εκεί που κάθεστε. Ευχαριστώ. Τον λοιπόν, καλό να έρθει να κάτσει δίπλα μου. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε την τροπολογία 15, άρχεται η ψηφοφορία. Πε, πέρας. Και εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. Άρχες ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 ελέγχουμε την 64 άρχεται η ψηφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1.14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές δεν σηκώσατε χέρι οπότε θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο της ψηφοφορίας άρχεται πέρας Ναι, εγκρίνεται. Ε, μου φέρνουν την ε, κάρτα ψηφορίας. Ε, είμαι υπέρ. Εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα 40 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 144 Πέρας. Εκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές πράσινη εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα τελική ψήφος, άρχιτη ψηφορία. And it is closed. Πέρας. Και εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ε, για την ε, θέσπιση προγράμματο για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ε, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Σημαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 πολλές μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 93 υπέρ κατά αποχές το γεφτητή έλεγχος για την 93 πέρας εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές. Η άλλη είναι υπέρ, όλη η ομάδα, ότι εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 101 πέρας εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 102 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σε τμήματα για την 103. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές η άλλη είναι κατά ή υπέρ. Έλεγχος τότε. Άρχεται η υπερ ελεγχο τοτε Πέρας. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές έλεγχος πέρας Ισοψηφία και απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κατά τμήματα 20. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Δεν ψηφίζουμε. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές. Το ECR εγκρίνεται. Ας γίνει έλεγχος όμως. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 33 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές δεν είδα τα χέρια 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά τμήματα η 61 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Τώρα ψηφίζουμε σχέδιο ψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Έτος Πρασίνων Πόλεων, πιο πράσινων πόλεων. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά, αποχές. Η πράσινη είστε υπέρ ή κατά. Ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 71. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά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 εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20 και 1 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30, μια προσθήκη. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχέ. Οι σοσιαλιστές είναι κατά, υπέρ, άρα εγκρίνεται. Συμβαστική 6, ποιο είναι υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 7, υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 49 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 50 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 50 άρχεται η ψηφοφορία Τώρα πράσινοι με μπέρδεψαν και οι φιλελεύθεροι. Μάλλον μεταξύ τους μπερδεύτηκαν. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. «51. Ποιος είναι υπέρ» κατά αποχές απορρίπτεται. «52. Υπέρ» κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «58. Υπέρ» κατά αποχές απορρίπτεται. Μία προφορική τροπολογία για την 56. Είναι κανείς κατά της προφορικής. Όχι, οπότε ψηφίζουμε την 56 με την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59. Ή μάλλον 57. 57 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και 60 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 60. Τέλος. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες, δεν έχουμε άλλες ψηφοφορίες για σήμερα. Περνάμε σε θέματα προσυζήτηση. Σας δίνω δύο λεπτά για να αποφασίσετε αν θα παραμείνετε ή θα αποχωρήσετε. Uh, Okay, if you wanna take your seats, the... Παρακαλώ, καθίστε. Παρακαλώ, καθίστε. Όσοι θέλουν να κάτσουν, οι υπόλοιποι μπορούν να συνεχίσουν τα πηγαδάκια τους έξω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κυρίες μου. Um, Ωραία τώρα. Ναι, θέσμιση κανονών για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ ε, και ε, η είναι ο κύριος Λαβία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την 1η Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση περί κανονισμού για τα στατικά σχέδια της κοινή ερωτικής πολιτικής που ουσιαστικά συναθρίζει τους δύο πυλώνες και τους ενώνει σε ένα κερματικό μέσο. Η τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει ένα νέο μοντέλο που βασίζεται επί νέων στόχων, τονίζοντας τους στόχους των πολιτικών για το περιβάλλον και για την αλλαγή του κλίματος είναι από τις νέους στόχους, τρεις είναι συγκεκριμένοι ειδικοί στόχοι που μπαίνουν στα πλαίσια της εντολής που έχει η Επιτροπή μας. Μείωση και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος με άλλα λόγια, να ευνοήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και να συμβάλλουμε έτσι την προστασία της βιοπικιλικότητας και να προωθήσουμε την οικονομία και να βελτιώσουμε την απάντηση που δίνει η γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της απαιτήσει τη κοινωνίας για υγιεινά τρόφιμα, συμπραγμένων ασφαλών, ε, βιωσίμων τροφίμων ε, και επίσης να προστατεύσουμε και τα ζώα, την ευημερία των ζώων. Πάνω σε αυτό το χαρτοφυλάκιο ζητήσαμε στη διάσκεψη των Προέδρων να είμαστε συνδεμένοι στις εργασίες επιτροπή και επισκευαζόμεθα βάσει του... Το άρθρο Κινούμεθα βάσει του 54. Έχουμε κοινή αρμοδιότητα για διάφορα άρθρα. Και εκεί επικέντρωσα εγώ την προσπάθειά μου και τις εργασίες μου και θα ήθελα να δώσετε προσοχή διότι είναι αυτά τα άρθρα που αφορούν την αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Επιτρέψτε μου πριν πω στην ουσία να αναφερθώ στο άρθρο 54 που θεωρητικά δίνει σε εμά κοινή αρμοδιότητα, αλλά στην πραγματικότητα η Επιτροπή Γεωργίας δεν μας την εκχωρεί. Δεν συμμετείχαμε, δεν προσκληθήκαμε στην ακρόαση της Επιτροπής, στο εργαστήριο της Επιτροπής. Δεν είχαμε κανένα ρόλο όσον αφορά τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος που δυνάμει του ε, άρθρου 54 από κοινού να καθοριστεί. Πήραν πληροφορίες μετά από τις αποφάσεις άτυπα Κάτι που προφανώς με οδηγεί να υπογραμμίσω και να το σημειώσω σαν γεγονός και μετά από μια συνάντηση με τους συντονιστές γράψαμε μια επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και στη διάσκεψη των προέδρων για να ληφθούν υπόψη όλα αυτά που συνέβησαν. Και τώρα προφανώς θα ήθελα να μπω στο θέμα μας. Είναι προφανές ότι σε αυτή τη θητεία έγιναν μια σειρά από τροποποίησεις στην ε, ισχύουσα νομοθεσία και κυρίως μέσω του κανονισμού Omnibus έγιναν διάφορες αλλαγές. Κατά την άποψή μου σίγουρα ε, βελτιώθηκε η νομοθεσία ε, και πρόσφατα μπήκαν αυτές οι αλλαγές σε ισχύ. Η ΚΑΠ είναι μία από τις ιστορικές θεμελιώδεις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η μόνη πραγματική κοινή πολιτική. Και είναι εξίσου σαφές ότι όπως ε, το συζήτησα μέχρι στην Ολομέλεια, στην ΚΑΠ θα πρέπει να, δοθεί, ε, να δοθούν επαρκείς πόροι ούτω ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρα τη κοινοτική πολιτική. Γι' αυτό επαναλαμβάνω τη σημασία που διατηρεί η ΚΑΠ ε, στον προπολογισμό χρειάζεται να έχει επαρκή προπολογισμό στο επόμενο δημοσιονομικό ε, πλαίσιο, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να γίνουν περικοπές γιατί έτσι θα αποδυναμωθεί η πολιτική. Απ' την άλλη πλευρά επιτρέψτε μου να αναφερθώ ε, στη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πλευράς γενικής αρχιτεκτονικής της. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που πάντα έλεγε ότι η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να είναι και να κρατήσει τον, το χαρακτήρα κοινοτικής πολιτικής. Σε κάποιους ε, δεν αρέσει ο διαχωρισμός, ε, δεν είναι καλή, καλός διαχωρισμός της κοινή πολιτικής σε 27 ξεχωριστές εθνικές πολιτικές. Καλή επικουρικότητα, δηλαδή τηρήσουμε το χαρακτήρα των κοινών της πολιτικής, θα έχουμε 27 διαφορετικές αγροτικές πολιτικές και προφανώς θα χάσουμε αυτό το χαρακτήρα της κοινή πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, κατανοώ ότι στο Συμβούλιο ο υπουργός που θα ε, αναλάβει το, τους πόρους και βάσει επικουρικότητας θα χειριστεί τους πόρους, ε, ποιος θα έλεγε όχι άμα έχει στρατηγικό σχέδιο και του δοθούν τα χρήματα. Εμείς το Κοινοβούλιο όμως πρέπει να διατηρήσουμε ε, την προσέγγιση της κοινοτικής πολιτικής όσον αφορά την ΚΑΠ. Και πάω τώρα στις διάφορες συγκεκριμένες προτάσεις. Οι προτάσεις μου συνδέονται σημαντικά με τις 52 τροπολογίες που υπέβαλα και, και αφορά περισσότερο η προσέγγιση μου τις περιβαλλοντικές πτυχές. Δεν ήθελα ε, στην έκθεση αυτή να σταθώ στα γενικά ζητήματα. Γι' αυτά προφανώς συνεργασία με άλλους συναδέλφους στην Επιτροπή Γεωργίας έχω υποβάλει τροπολογίες στα πλαίσια εκείνου του πλαισίου. Οι 52 τροπολογίες ουσιαστικά φορούν τα άρθρα της κοινή αρμοδιότητας των Επιτροπών. Πιο συγκεκριμένα, τροποποίησε τη διατύπωση δύο των, από τους δύο στόχους, νέους στόχους, να γίνουν πιο συνεκτικοί, να ταιριάσουν καλύτερα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Στάθηκα στο κείμενο όσον αφορά την αρχιτεκτονική, το New Delivery Model που βασίζεται στους στατικικούς εθνικούς πυλώνες, σαφώς έκανα κάποια αναφορά στην αιρεσιμότητα ε, και θα σταθώ σε αυτά τα στοιχεία αργότερα. Ε, δέχτηκα θετικά το νέο ενισχυμένο διευρυμένο σύστημα της αιρεσιμότητας και το οικολογικό υποχρεωτικό σύστημα ε, που θα είναι για τα κράτη-μέλη θελοντικό για τους γεωργούς και μπορεί να αποζημιώσει τους γεωργούς που συγκεκριμένα συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματολογικών περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους εθνικούς στόχους Πιστεύω ότι η νέα πρόταση αφήνει μεγάλη διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη όσον αφορά τη δαπάνη των πόρων και τον καθορισμό σε επίπεδο φιλοδοξιών. Από τη στιγμή που αυτό θα μπορούσε δυστυχώ να οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα χαρακτηρίζεται και από αυτή την άποψη από 27 διαφορετικέ πολιτικέ με φιλοδοξίε διαφορετικέ, και έτσι θα χάσουμε την κοινή ψυχή τη ΚΑΠ. Θα, εγώ ήθελα τι κοινέ πτυχέ προτάσεω να στηρίξω βάζοντας στη βασική πράξη κάποια στοιχεία που η πρόταση άφηνε στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών, μειώνοντας ακριβώς ε, την εθνική προσέγγιση για να τονίσω περισσότερο τον κοινοτικό χαρακτήρα. Βέβαια, είναι θετική μεγαλύτερη ευελιξία βάσει τη επικουρικότητα, αλλά εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν αποκλίνουσε προσεγγίσει, αντιμετωπίζοντα του γεωργού με τρόπου εντελώ διαφορετικά όταν έχουν παρόμοια δραστηριότητα και κάνουν ίδια εργασία. Ενίσχυσα λοιπόν τα κοινά στοιχεία της κοινή ερωτική πολιτικής. Γι' αυτό πρόσθετα κάποια ε, στοιχεία στη βασική διάταξη, μικρώνοντας την διακριτική ευχέρεια, να μην έχουμε επανεθνικοποίηση της πολιτικής. Αλλά υπάρχει ευελιξία στην τροπολογία 18, προβλέπω ότι τα κράτη-μέλη στην τροπολογία 18 που προβλέπει τα κράτη-μέλη θα καθορίζουν τον κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που είναι ευεργετικές για το κλίμα και το περιβάλλον ε, και ουσιαστικά το άλλαξε αυτό με τέτοιο τρόπο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτει μια κατεξοδότηση πράξη που καθορίζει τον κατάλογο και τις πρακτικές τις γεωργικές που είναι καλές για το περιβάλλον και για το κλίμα και μπορούν μέσω των πρακτικών αυτών τα κράτη-μέλη να επιλέξουν εκείνες από εκείνε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει στην κατεξοδότηση πράξη, ούτω ώστε να τηρήσουμε τον κοινοτικό χαρακτήρα και να αφήσουμε όμω και μια δυνατότητα επιλογή στα κράτη-μέλη. Ε, παρουσιάσε και κάποιε τροπολογίε που προβλέπουν την αύξηση του αριθμού των στόχων και παρεμβάσεων που το κράτο μέλο θα πρέπει να εφαρμόσει σε διάφορου τομεί, ενισχύοντα λοιπόν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα τη πολιτική και αυξάνοντα έτσι το περιθώριο παρεμβάσεω των ίσων παρεμβάσεων που θα πρέπει να βάλουν στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο τα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι η προσέγγιση τη προτάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώ προσανατολίζεται προ τα αποτελέσματα και αυτό απαιτεί ένα στέρεο πλάσιο που θα επιτρέπει μια αξιολόγηση και έναν έλεγχο που θα είναι επαρκή για την δώσει αποτελέσματα πολιτική σε σχέση με συγκεκριμένου στόχου που έχουν καθοριστεί σε κάθε κράτο μέλο. Σε αυτό το εγχείρημα θα πρέπει να προσέξουμε πολύ, να αποφύγουμε διάφορα κενά και να εγγυηθούμε μια ε, ευθύνη όσον αφορά τις δαπάνες και τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τους ορισμούς, σε κάποιες περιπτώσεις εγώ αναφέρθηκα σε αυτό που μεγάλη δυσκολία και με μεγάλη διαδικασία επετεύχθη εντός των πλαισίων του κανονισμού Omnibus, αποφεύγοντας έτσι μετά από δύο χρόνια του Omnibus ε, να αλλάξουμε ε, πορεία. Διότι η συμφωνία που επετεύχθη θεωρούσα τότε ότι ήταν πολύ ε, τη συμφωνία από αυτά που πρότεινε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαφές ότι έκανα και προτάσεις όσον αφορά τους νέους, όσον αφορά την ευελιξία για τις μεταφορές. Έδωσε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις αρχές διαχείρισης. Προφανώς ε, και σε σχέση με όλα τα κράτη-μέλη που έχουν περιφερειακές αρχές ε, διαχείρισης και όχι εθνικές, δίνοντας τη δυνατότητα δυνατότητες να μην αλλάξουν κατεύθυνση για να συμμορφωθούν παρενέβη μετά στο θέμα της θέσης σε ισχύ. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα που ανήκει αποκριστικά σε εμά, αλλά και από αυτού θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε. Πιστεύω να εκφράσουμε άποψη. Στην προηγούμενη θητεία ήμουν εισηγητή του οριζόντιου κανονισμού για την ΚΑΠ και κάναμε πολλού τριμερεί διαλόγους για να καθορίσουμε στο, καταλήξουμε στον ορισμό. Εάν πάνε τα πράγματα καλά, θα φτάσουμε σε ψηφοφορία στην πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια και βλέποντας τις επικείμενες ε, ευρωεκλογέ, τη διαμόρφωση νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη δημιουργία του νέου Κοινοβουλίου και την αδυναμία να ξεκινήσουμε αμέσως τους τριμερείς διαλόγους και λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των τριμερών διαλόγων που κατά το παρελθόν ήταν αναγκαίοι για να καθαρίσουμε σε ένα καθορισμό πολιτικής που είναι τόσο σημαντική, πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο 2020 για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και δεν πιστεύω ότι πρώτη Ιανουαρίου του 2021 μπορεί να μπει σε εφαρμογή νέα πολιτική. Γι' αυτό πρότεινα μια αναβολή τη ισχύω τη νέα πολιτική, διατηρώντας αυτό που είχε καθοριστεί στα πλαίσια του κανονισμού Omnibus. Και θα κλείσω εδώ λέγοντας ότι όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση γνωρίζουμε πολύ καλά και ποιος είναι ο σημαντικός αριθμός των τροπολογιών που κατέφτασαν βάσει της προτάσεως αυτής στην Επιτροπή Γεωργίας. Είναι αρκετές οι τροπολογίες. 4.408 δεν είναι ε, μικρός αριθμός. Οπότε αυτό δυσχεραίνει έτσι περαιτέρω τη διαδρομή από τώρα μέχρι τη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Και θα ήθελα και οι δύο επιτροπές, όπως προβλέπετε στο άρθρο 54, να μπορέσουν να επεξεργαστούν το υλικό των αρμοδιοτήτων μας με κοινή αρμοδιότητα και να μην γίνει προσπάθεια από την Επιτροπή Γεωργίας να επικρατήσει ε, επί των δικών μας νομοδοτήσεων που θα πρέπει ψηφιστούν. Ε, θα πρέπει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας, να λάβουμε υπόψη και αυτό που θα αποφασιστεί στην Επιτροπή Γεωργίας, ούτως ώστε η δική μας ψηφοφορία να γίνει εν ευθέτω χρόνο και μετά αυτό που θα αποφασίσουμε η Επιτροπή Γεωργίας να μπορεί να το δει και να τοποθετηθεί. Και εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα στρέφουμε προς τους ε, σκιώδεις, όμως ε, θα πρέπει να είμαι αυστηρή ε, όσον αφορά το χρόνο σας, όχι περισσότερα λοιπόν από τρία λεπτά. Η κυρία Μελιόρα αρχικά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη διότι θα αναφερθώ σε μερικά σημεία μονάχα. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Ε, με την αξιολόγηση σχετικά με τα τρία σημεία ότι εδώ πέρα θα χρειαζόμαστε περισσότερο ευρωπαϊκή πολιτική και όχι εθνικοποίηση. Το δεύτερο σχόλιο στο οποίο συμφωνώ απολύτως είναι τα όσα είπε για την ε, διαδικασία και εκεί είμαι ε, κάπως σκεπτικιστική και το τρίτο σημείο το οποίο πραγματικά υπογραμμίζω είναι η μεταφορά των μέσων με τον ε, τρόπο που ε, προτάθηκαν είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε και εμείς στο S&D. Είναι κάποια θέματα τα οποία θα φανούν όμως και στις τροπολογίες μου. Αρχικά το ερώτημα της ε, σύνδεσης των σκοπών και εδώ θα έχω κάποιες τροπολογίες. Αυτό θα πρέπει να είναι εφικτό και στον πρώτο αλλά και στον δεύτερο πυλώνα και αυτό το οποίο μπορεί να συνεισφέρει η Επιτροπή Envy είναι να έχουμε χρήματα από τον μεγάλο κορβανά της ε, ε, ΚΑΠ για τους κλιματικούς στόχους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θα πρότεινα λοιπόν ε, στον δεύτερο πυλώνα από το 50% των ποσών αυτών να φαίνεται ξεκάθαρα. Επίσης, στόχος θα πρέπει να είναι όχι μονάχα τα κλιματικά ζητήματα, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα θα ήθελα να υπενθυμίσω ε, εκθέσεις από το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο μας είπε ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να ε, έχουν συγκεκριμένους ε, στόχους, να χρησιμοποιούνται για την βιοπικιλότητα, να κάνουμε περισσότερα για το κλίμα. Τώρα όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τον διαχειρισμό αυτών και εκεί είμαι σκεπτικιστική, δεν είναι καλό το πώς, το πώς παρουσιάζεται για το κλίμα διότι προωθεί ιδιαίτερο. στον το ε, τομέα κρέατος ε, και ε, θα μπορούσαν αυτά να χρηματοδοτηθούν και από άλλα μέσα χωρίς ε, να χρειάζονται περαιτέρω συνδεδεμένες πληρωμές. Επίσης, ε, η ερησιμότητα θα πρέπει να ενισχυθεί, όλες οι άμεσες πληρωμές ε, θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το οποίο σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι αγρότες να κάνουν περισσότερα, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί για την προστασία του περιβάλλοντος, να χρησιμοποιούν, μειώνουν μάλλον τη χρήση ε, ζυζανιοκτώνων ε, και να συνεισφέρουν ε, ως προς την προστασία του εδάφους και του κλίματος γενικότερα. Στο άρθρο 6 λοιπόν θα πρέπει αυτό να γίνει πιο ξεκάθαρο. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι ε, οργανισμοί για την προστασία του ε, ε, περιβάλλοντος ε, αλλά και ε, επιστήμονες λένε ότι δεν κάνουμε αρκετά για το περιβάλλον οπότε θα πρέπει να είναι μεν εθελοντικό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο συνολικό για τα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε τους νέους αγρότες και τα προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι τροπολογίες λοιπόν δεν θα είναι συνολικά 4.000, όμως θα αφορούν σίγουρα τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία θέλουμε να τονίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για την πολύ καλή του έκθεση με το νέο μοντέλο της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, νιώθω ανάμεικτα συναισθήματα. Παρόλο που σε πολλά σημεία συμφωνώ με τον εισηγητό. Απ' τη μια χαίρομαι που εκχωρούνται περισσότερες αρμοδιότητες πια στα κράτη-μέλη, κάτι που θα οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση των κονδύλιων. Απ' την άλλη όμως φοβούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ε, διοικητικές επιβαρύνσεις και διατυπώσεις και γραφειοκρατία και οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες αρχές. Γι' αυτό θα ήθελα να δηλώσω την υποστήριξή μου ε, για την τροπολογία του εισηγητού που προτείνει μια αναβολή για την εφαρμογή του νέου μοντέλου. Επίσης, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το, τουλάχιστον το ισχύον επίπεδο χρηματοδότησης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Φοβούμε όμως ε, ότι θα ε, διευρυνθεί το πεδίο των στόχων ε, των κλιματικών και των περιβαλλοντικών. Σίγουρα και η Γεωργία θα πρέπει να συμβάλλει στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και στο περιορισμό των εκπομπών του θερμοκηπίου. Φοβάμαι όμω ότι οι διοικητικέ επιβαρύνσει που θα προκύψουν από τέτοια περιβαλλοντικά κριτήρια ίσω ε, έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Για, από την δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε με υπερβολικές διοικητικέ διατυπώσεις του γεωργού, που στόχο έχουν κυρίως στην παραγωγή ε, υγιεινών και ποιοτικών τροφίμων. Επίσης, ε, είμαι κατά των υπερβολικών επιβαρύνσεων λόγω κλιματικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, γιατί κάτι τέτοιο ίσως διαταράξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργών στι παγκόσμίε αγορέ. Και σίγουρα οι γεωργοί των ε, λιγότερο εύπορων χωρών ε, δεν θα έχουν την αρκετή χρηματοδότηση για να προσαρμοστούν ε, στη μετάβαση αυτή. Οπότε τα στρατηγικά σχέδια για να ευοδοθούν θα πρέπει να τη χάνουν τις κατάλληλες χρηματοδότησης. Γι' αυτό και θα καταθέσω τροπολογίες για την εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων για τους γεωργούς και την μεγαλύτερη ελαστικότητα στις μεταφορές κονδυλίων μεταξύ των δύο πυλώνων. Δεν συμφωνώ με τον εισηγητή που προσπαθεί να περιορίσει αυτή την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων. Επίσης, ε, ε, το εύρος των κατεξοδότηση πράξεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερβολικά μεγάλο. Σε μερικές περιπτώσεις το περιορίζει αυτό ο εισηγητής, αλλά φοβάμαι ότι ε, έτσι θα προσταθούν οι δείκτες που προβλέπονται στο άρθρο 7. Οπότε οι τροπολογίες μου θα έχουν στόχο να περιορίσουν αυτές τις εξουσίες της ε, Επιτροπής. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κερμπράντη. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. συμφωνώ και υποστηρίζω την, το σχέδιο ε, του Τζοβάνι. Θα ήθελα να ε, ξεκινήσω λέγοντας ότι όσον αφορά τα περιβαλλοντικά σημεία τα οποία αναφέρει έχει απόλυτο δίκιο. Πριν όμως ε, περάσω στο πρασίνισμα ε, και στον πυρήνα του δικού μας ρόλου σε όλη αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα προς την Επιτροπή. Γνωρίζουμε ε, λοιπόν ότι η Επιτροπή έχει έναν οργανισμό ε, που ε, βασίζεται στα δεδομένα, όμως με κάποιο τρόπο εδώ πέρα χάνεται η κάθε λογική. Δεν υπάρχει καμία λογική στην πρόταση, είναι καθαρά πολιτική και δεν βασίζεται στα δεδομένα. Ευτυχώ όμω ε, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο σε δύο αυστηρέ εκθέσεις του, τον Απρίλιο και στις 7 Νοεμβρίου η δεύτερη, μας έδειξε το πόσο έντονο είναι, το, είναι η έλλειψη λογικής ε, στην ε, πρόταση της Επιτροπής. Πρώτον βασίζει την πρότασή της στο γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί κλειδί για την αγροτική οικονομία δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο διότι ε, κυριαρχείται από τη βιομηχανία ε, και τις υπηρεσίες. Ο ε, αγροτικός τομέας μαζί με την αλληλεία αντιστοιχεί μόλις το 4% της συνολικής οικονομίας των αγροτικών περιοχών. Επίσης η οδηγία για, τις, για την άμεση υποστήριξη έρχεται από το ίδιο το αγρόκτημα. Στην συνέχεια όλα τα επιπρόσθετα δεν συνυπολογίζονται στη συγκεκριμένη οδηγία, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ελάχιστα ε, εισοδήματα από τα αγροκτήματα, διότι αν κάποιος εργάζεται κάποιο, κάπου αλλού και αυτό δεν συνυπολογίζεται στα δεδομένα για την οικογένεια, τότε φυσικά και λαμβάνεις μεγαλύτερη υποστήριξη. Η λογική λοιπόν πίσω από την ε, πρόταση αυτή δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα την απάντηση της Επιτροπής ε, σε αυτή την κριτική ε, που ασκείται από την πλευρά του ελεκτικού συνεδρίου. Τώρα όσον αφορά το πρασίνισμα, συμφωνώ ε, με τον ε, Τζοβάνι ότι αυτή η λογική θα ήταν επικίνδυνη αν δεν είχαμε ένα σύστημα ούτω ώστε τα μέτρα αυτά να αντικατοπτρίζονται σε εθνικές πολιτικές, διότι γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ένα και μόνο συμφέρον όσον αφορά την ΚΑΠ, το οποίο είναι να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για τα αγροκτήματά τους τα κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται για τα κριτήρια πρασινίσματος τα οποία θέτουμε και ας λοιπόν ας είμαστε ειλικρινείς. Ούτε το ίδιο συμβαίνει και με το Κοινοβούλιο εδώ πέρα. Την τελευταία φορά το, ε, η Επιτροπή Άγκρη απέρριψε όλες τις προτάσεις προ, ε, πρασινίσματος από την Επιτροπή. Οπότε η Επιτροπή είναι η μόνη, ο μόνος θεσμός που υπερασπίζεται το περιβάλλον και είναι μόνοι τους εδώ πέρα σχετικά με την πρότασή τους. Θα Έχουμε μια ισχυρή ε, απέτηση λοιπόν έχουμε μετρήσιμους στόχους βιωσιμότητας στην πρόταση ΚΑΠ και αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι εν τέλει ο αγροτικός τομέας θα παίξει τον ρόλο του στην βιώσιμη οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Έικαουτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάντοτε είναι δύσκολο να μιλήσεις μετά από τον Γιάννη διότι και εγώ ε, θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενος ε, στο ελεγκτικό συνέδριο, όμως ε, τελικά δεν μπορώ να το κάνω, μου στέρισε αυτή την ευκαιρία ο Χέρμεν Γιάνν. Όμως παρόλα αυτά θα ήθελα να ακούσω από την Επιτροπή το Πώ θα απαντήσουν στα όσα είπε το ελεκτικό συνέδριο, διότι αυτά τα οποία ισχυρίζονται είναι πολύ σοβαρά. Και θα ήθελα να τονίσω ε, κάποια θέματα τα οποία ε, σχολιάσουν στην αξιολόγηση αντικτύπων. Ε, πρώτον, ε, όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις ε, δεν υπάρχει καμία αναφορά εκεί. Ε, την επιβολή χρήσης αυτών με βάση τα εκτάρια εδάφους και ότι αυτό δεν είναι αντίστοιχο για την αντιμετώπιση ανησυχιών για το περιβάλλοντος. Όλα αυτά φαίνονται μη ρεαλιστικά παρά τις φιλοδοξίες της Επιτροπής ε, η πρόταση φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία φιλοδοξία για το περιβάλλον. Φαίνεται ότι η Επιτροπή ε, στρέφεται προς μια απόδοση χωρίς όμως να παρουσιάζει ένα αποδοτικό σύστημα ε, και είναι δύσκολο το πώς θα καταλάβουν, πώς θα το επιτύχει αυτό η Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Ως πράσινος ε, θα λέγατε ότι είναι αναμενόμενο να το πει αυτό. Όμως τώρα να γυρίζει και να λέει το ελληνικό συνέδριο ότι η Επιτροπή δεν κάνει καλή δουλειά, αυτό είναι σοβαρό και εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να το πάρουμε ε, σοβαρά. Αν θέλουμε μια ΚΑΠ που να αποδίδει καλύτερα και για το περιβάλλον, τότε θα πρέπει να ε, ζητήσουμε μεταρρύθμιση των όσων προτείνει η Επιτροπή και θα ήθελα να συγχαρώ τον Τζοβάνι διότι στο έργο του λέει, το αναφέρει αυτό. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί. Πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή έτσι όπως το θέτεις, όμως ως πράσινος θα σε βοηθήσω να το ισχυροποιήσει το κείμενο. Ακούμε το ελεγκτικό συνέδριο, συνέδριο και από πλευρά τη Επιτροπή θα ήθελα να ακούσω το πώ θα αντιδράσουν σε αυτό και πώ θα προσαρμόσουν τι προτάσει αυτέ, διότι μπορείτε να το κάνετε. Θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα ε, μείνετε κολλημένοι στο κείμενό σας και στις προτάσεις, θα πείτε αυτή είναι η πρότασή μας και θα την υπηρεσπιστούμε ή θα λάβετε υπόψη σας ε, αυτή την κριτική από ένα σοβαρό θεσμό και θα ε, προσαρμόσετε αναλόγως τις προτάσεις σας όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σίγουρα θα ε, το συζητήσουμε ε, με τον εισηγητή και ελπίζω αυτή τη φορά έτσι για αλλαχή η Άγκρη θα αρχίσει να μας ακούει παρά να λέει ότι είναι χρήματα αγροτών. Είναι χρήματα φορολογουμένων και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα φορολογουμένων χρησιμοποιούνται ορθά και θα το διασφαλίσουμε αυτό και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα μας βοηθήσει ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρότασή τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ικχάουτ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο κατάλογος των σκιωδών και πάμε στα μέλη που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Αρκετοί είναι στον κατάλογο. Θα θέσουμε όριο χρονικό. Δίλεπτο. Παρακαλώ να το τηρήσετε. Οι δεμή θα χάσουμε τον έλεγχο. Θα βγούμε εκτός προγράμματος. Ο κ. Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σωστά τα είπε ο Τζοβάνι Λαβία. Στη δουλειά που κάνουμε εδώ στην ΕΜΒΗ θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί των δικών μας αρμοδιοτήτων. Αυτό δεν ισχύει μόνο για αυτό το χαρτοφυλάκιο, αλλά και άλλα δύο. υπάρχει και αλλού ε, πρόβλημα αρμοδιοτήτων. Πιστεύω ότι ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει μια κοινή πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο το New Delivery Model πρέπει να το προσέξουμε. Να παραμείνει ο κοινωτικός χαρακτήρας. Ε, εδώ στις πολιτικές που συζητούμε, βιωσιμότητας, ίσως χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση σε διάφορα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε πιο πράσινη αγροτική πολιτική που σέβεται το περιβάλλον και να είναι βιώσιμη. Ίσως να υπάρχει και εθνική και περιφερειακή αρμοδιότητα γι' αυτό. Να λαμβάνονται υπόψη συνθήκες εργασίας που ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Οι γεωργοί δεν είναι αρνητική όσον αφορά βιωσιμότητα. Πρέπει να αλλάξουμε εμεί τη διατύπωση. Στην αγροτική πολιτική δίνουμε την εντύπωση ότι κρατάμε τα χρήματα και αν δεν γίνει πιο πράσινη γεωργία δεν τα απελευθερώνουμε. Δεν είναι σωστή προσέγγιση. Θέλουμε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Και αυτό γίνεται μόνο με βιώσιμη γεωργία. Η βιωσιμότητα είναι κομμάτι της ποιότητας. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς το αφήγημά μας. Να έχουμε κανόνες κοινά αποδεκτούς, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. δεν κατάλαβαν καλά την έννοια του πρασινίσματος η Γεωργοί, γιατί είναι μια κάπως παράλογη έννοια όπως την παρουσιάζουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητε διαφόρων περιοχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γίνει πιο βιώσιμη η γεωργία. Δεν το κατανόησαν οι γεωργοί. Το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι η η προσέγγιση μα μέχρι τώρα. Πρέπει οι κανόνε μα να γίνονται κοινά αποδεκτοί. Και αν το κάνουμε αυτό θα είναι, θα είναι με το μέρο μα και η Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ντελαή έχει το λόγο δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ χαιρετίζω το έργο του συναδέλφου μας, του κυρίου Λαβία. Έχω κάποια απορία σε αυτά που έλεγε για το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να πω ότι δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε και τη δική μας νομοδότηση λόγω χρονοδιαγράμματος. Τον υποστηρίζω όσον αφορά τις γενικές απόψεις, ε, η θέση ισχύει το 2023, ότι ε, το άρθρο 6 στόχοι πρέπει να βελτιωθούν, η καινοτομία του άρθρου 43 επίσης πρέπει να τονιστεί. Έχω κάποια σχόλια στη, όσον αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στου στόχου 8 και 9, τι αναφέρει. Πρέπει να προωθήσουμε απασχόληση στην ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη, την τοπική, στην ύπεθρο και τη βιολογική οικονομία και την, την ε, υλοτομία την βιώσιμη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση όμω. Θα ήταν εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ένα σχέδιο ε, πρωτεϊνών που θα ενταχθεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο στα πλαίσια της ΚΑΠ. 70% των φυτικών πρωτεϊνών εισάγουμε και προέρχεται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αυτή. Και δεν, θα έχουμε, δεν έχουμε αυτονομία διατροφική πάνω σε αυτό. Η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να έχει φιλόδοξους στόχους, οικονομική επίδοση σωστή και περιβαλλοντική να έχει, για να μην υπάρχει αντίθεση πλέον μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος. Προστασία του περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να αποτελεί περιορισμό για τη γεωργία. Πιστεύω αντίθετα ότι είναι ένα πλεονέκτημα πραγματικό για τη γεωργία, για μια γεωργία που είναι υπεύθυνη. Όπως είπε και ο συνάδελφος Ντόρφμαν, η αιρεσιμότητα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψει στο θα πρέπει να, ε, να, μην είναι, να εφαρμόζει μέτρα σωστά μένα, αλλά να μην είναι οικονομικά βιώσιμο. Λοιπόν, θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίε να τα διορθώσω αυτά τα στοιχεία. Κυρία Σράιρ Πίρικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας τον κύριο Λαβία. Συμφωνώ με τις προτάσεις του και συμφωνώ και με τον κύριο Ντόρφμαν, οπότε δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα σχόλιά τους. Ε, σίγουρα, αν θέλουμε να συμβιβάσουμε και να συνδυάσουμε τη γεωργία με τη φύση, θα πρέπει να συνεργαστούν οι δύο, οι δύο επιτροπές, γεωργίες και περιβάλλοντος. Θα πρέπει οι δύο επιτροπές ε, να συνεργαστούν για να καταλήξουν σε κοινό αποτέλεσμα. Ο κύριος ε, Κερμπράντι έκανε κάποιε παρατηρήσει με τις οποίες δεν συμφωνώ απόλυτα. Στην Ολλανδία έχουμε 168 περιοχές του Natura ε, και χιλιάδες γεωργοί συμμετέχουν σε αυτές. Φυσικά είναι διαφορετικοί περιορισμοί. Επίσης έχουμε το 30% στους πυλώνες και τη δυνατότητα επιβράβευσης των γεωργών για τις προσπάθειές τους αντί να τους περιορίζουμε ακόμη περισσότερο ή να τους επιβαρύνουμε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά σημεία και ελπίζω να καταλήξουμε τελικά. Γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τα γεωργικά εισοδήματα, γιατί αν δούμε και το θέμα της ασφάλειας τροφίμων και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, δεν είναι προφανή όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν αρκετά κονδύλια και να φτάνουν στους γεωργούς, τους άμεσα δικαιούχους. Και κύριε Γερμπράντη, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να φτάνουν τα χρήματα στα σωστά χέρια. Και αν μιλούμε μόνο για κονδύλια για την καινοτομία της αγοράς, δεν αρκεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει τα χρήματα να φτάνουν στους γεωργούς τους ίδιους. Και επίσης να φροντίσουμε να υπάρχουν επαρκή κονδύλια και για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης. Ευχαριστώ. Κύριε Αγιούσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Λαβία για την πρότασή του και να πω ότι σε γενικέ γραμμές συμφωνώ με τον εισηγητή μα και κυρίω σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του επίπεδου χρηματοδότηση τη κοινή γεωργική πολιτική. Είναι σημαντικό να παραμείνει αλόβητο ο γεωργικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, να αποφύγουμε τη διακριτική ευχαίρεια που δίνει, την υπερβολική διακριτική ευχαίρεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Θα, δεν θα πρέπει να υποπέσουμε στο σφάλμα να έχουμε 27 διαφορετικέ γεωργικέ πολιτικέ. Επίσης, συμφωνώ θα πρέπει να αναβληθεί η θέση εφαρμογής το 2023. Γιατί όχι μόνο είναι πολλές ε, οι αλλαγές, αλλά δεν μπορούμε σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να εφαρμόσουμε το νέο μοντέλο. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα ε, που εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ε, θα καταθέσω τροπολογίες στα άρθρα 5 και 6 που αφορούν τους στόχους και θα ήθελα να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη της εξασφάλισης της ε, επιστηστικής ασφάλειας και να αποφύγουμε την απερίμωση της υπαίθρου. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7, τους δείκτες, θα περιλάβω και νέους δείκτες με τις τροπολογίες για την ε, συμβολή των δασών ε, στην προστασία του περιβάλλοντος και την διέξοδο σε εξωτερικές αγορές. Επίσης, ε, να διαγραφεί η δυνατότητα να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω καταξιοδότηση πράξεων να προσθέτει νέους δείκτες. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 42 για τα απορροκυπευτικά, πιστεύω ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε το 10% των ε, λειτουργικών των επιχειρησιακών κονδύλιων που θα πρέπει υποχρεωτικά να πηγαίνουν σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τη μελισσοκομεία, να μπορούμε να αυξήσουμε από 50% σε 75% το ποσοστό χρηματοδότησης και επίσης ε, για τον κατάλογο των μέτρων που μπορούν να καλύπτονται από τα προγράμματα στήριξης πιστεύω θα πρέπει να συμπεριληφθεί και με λησοκομεία που έχει σημαντική περιβαλλοντική ε, προσφορά συμβολή. Και για τον Ίνο χρειαζόμαστε επενδύσεις και για την καινοτομία. Σε ό,τι αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του άρθρου 65 θα πρότεινα να είναι υποχρεωτικά αυτά τα μέτρα σε όλα τα κράτη-μέλη και οι ενισχύσεις ε, να δίνονται να καταβάλλονται όχι μόνο ως ε, αποζημίωση για γεωργό που εξέρχεται από την δραστηριότητα, αλλά να δίνονται και ως κίνητρο έναυσμα για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Γκροστέτ, ευχαριστώ. Δεν είχα την πρόθεση να παρέμβω στη συζήτηση γιατί την αλήθεια ότι τα θέματα της Επιτροπής Γεωργίας ε, δεν τα γνωρίζω τόσο καλά, αλλά μετά από την παρέμβαση του εισηγητού θα ήθελα να ζητήσω και εγώ το λόγο για να προσφέρω την αμέριστη υποστήριξή μου προς τον εισηγητή. Πραγματικά στενίζομαι πλήρως ε, το σχόλιο του και δεν πιστεύω ότι ε, τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας θα πρέπει να μονοπολούν μονίμως ε, τα θέματα της γεωργίας και να στερούν το λόγο από τις υπόλοιπες επιτροπές και κυρίως από τη δική μας. Δεν μου αρέσει ο όρος πρασίνισμα η οικολογικοποίηση της ε, γεωργίας. Προτιμώ να μιλούμε για βιώσιμη γεωργία, γιατί όταν μιλούμε για βιώσιμη γεωργία υπάρχει και κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική πτυχή και σίγουρα ο Γεωργός βρίσκεται στην καρδιά της κοινή γεωργικής πολιτικής και θα πρέπει να παραμείνει η ΚΑΠ η πιο σημαντική ε, ε, κοινοτική πολιτική. Και θα ήταν καταστροφή να επανέλθουμε σε μια επανεθνικοποίηση της γεωρικής πολιτικής. Ε, με εξέπληξε ο κύριος Ντόρφαν που μίλησε για απαιτήσει που δεν μπορούν να είναι ίδιε για όλε τι περιφέρειε. Ναι, το γνωρίζουμε αυτό. Οι αρχέ θα πρέπει να είναι οι ίδιε για όλου. Και φυσικά να τι προσαρμόζουμε στι ιδιαιτερότητε των περιφερειών. Γιατί έχουμε τι κλιματικέ αλλαγέ, τη χρήση των φυτοφαρμάκων που διαφέρει από ε, χώρα σε χώρα ή από περιφέρεια σε περιφέρεια. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα, αλλά οι αρχέ να είναι ίδιε για όλου. Και επίση ε, θα εξετάσω πολύ διεξοδικά αυτή την πρόταση και ίσω καταθέσω και τροπολογίε. Σας ευχαριστώ. Κύριος Χαϊταμα. Yes, thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγήτη για την έκθεση του. Έχω ε, μια παράκληση, μια προειδοποίηση να βελτιώσουμε ε, τα μέτρα για το πρασίνισμα. Όλοι συμφωνούν ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Το ελεγκτικό συνέδριο το λέει δεν αρέσει στους αγρότες, οπότε πραγματικά θα πρέπει να το ελάξουμε και αυτό. Το οποίο πιστεύω λοιπόν είναι ότι ο λόγος για τον οποίο δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή είναι επειδή βασίζονται στα μέτρα. Ως απρότης λοιπόν θα πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη προσέγγιση που σου, ορίζει, ε, που σου ορίζουν οι Βρυξέλλες, όμως εγώ δεν μπορώ να το κάνω ας πούμε στη φάρμα μου και το αποτέλεσμα. Οπότε απλά ε, τικάρουμε ορισμένα κουτάκια χωρίς να ε, κοιτάμε το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο αν θέλουμε να βελτιώσουμε το πρασίνισμα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια προσέγγιση με βάση το αποτέλεσμα που θα μπορεί να εκπληρωθεί με διάφορου τρόπου και έτσι υπάρχει δυνατότητα επιχειρηματικότητα για νέε ιδέε, καινοτομίε, ούτω ώστε οι αγρότε να συνεργαστούν, να συνεργαστούν ίσω και με άλλα ε, μέρη της επιστημιστικής αλυσίδας ε, και δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να είναι πολύ αυστηρή η διαδικασία, θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα και συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα αποτελέσματα σχετικά με τα, με το, με τα χρήματα που θα δαπανούνται και επίσης δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια ε, κρατική ότι φοβούμαστε την επανεθνικοποίηση οπότε να έχουμε πάλι ε, την προσέγγιση με βάση τα μέτρα. Μην το κάνετε διότι δεν θα λειτουργήσει. Επικεντρωθείτε στα αποτελέσματα, να έχετε ξεκαθαρούς στόχους εκεί, να αποτρέψετε την επανεθνικοποίηση ε, με τα καλά αποτελέσματα και θα πρέπει να θυμόμαστε, είναι να επικεντρωθούμε μονάχα στην πληρωμή με βάση το έδαφος. Όχι, θα πρέπει να έχουμε πληρωμές με βάση την δράση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάουσιλινγκ. Αυτό ε, όσον αφορά τη συνεργασία Άγκρη και NV συνάδελφοι της, ε, του ΕΛΚ θα πρέπει να ε, κοιτάξουν τον εαυτό τους ώστε να αποτραπεί αυτό. Γνωρίζετε ότι από την πλευρά των ε, συντηρητικών υπάρχουν ε, δισταγμοί όσον αφορά την ε, συνυπευθυνότητα της ΕΝΒΗ διότι χωρίς μία ορθή ΚΑΠ δεν πρόκειται να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους, τους στόχους βιωσιμότητας και βιοποικιλότητας. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό. Στην πρόταση της Επιτροπής τώρα θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή ε, εργάζεται ε, ωστόσο ώστε ε, να, ολοκληρωθεί, να τελειώσει την ΚΑΠ και να δημιουργήσει 27 διαφορετικές πολιτικές. Αυτό το οποίο με τρομάζει περισσότερο σε αυτή την πρόταση είναι ότι τα μέτρα για το περιβάλλον είναι εθελοντικά. Λέμε δηλαδή κάντε ό,τι νομίζετε εσείς ως ορθό έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη με τα χαμηλότερα ε, πρότυπα είναι αυτά τα οποία και θα ορίσουν την συνολική ταχύτητα. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να καθοριστούν οι πληρωμές με βάση την κλιματική πολιτική, με τους στόχους ε, ε, για το περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να πούμε ότι εσύ έχεις τόσα εδάφη, τόσες πληρωμές θα πάρεις. Αυτός είναι ο πιο ανόητος τρόπος να το προσεγγίσουμε. Θα πρέπει να έχουμε να επικεντρωθούμε στις εξαγωγές. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε τρεις στόχους και ο τελευταίος να είναι το περιβάλλον. Δεν είναι ορθή πολιτική ε, αυτή. Όταν ο κύριος Χόγγεν λοιπόν είπε ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν το πολύ κατάλαβε, τότε το βλέπω απαράδεκτο τρόπο να το πει αυτό, διότι προφανώς δεν ξέρει τι είναι σωστό. Οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε ούτως ώστε να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάνμπαχ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ είμαι ε, μέλος της Επιτροπής Ελέγχων των Υπολογισμών. Ε, και ε, ήμουν υπεύθυνη για οτιδήποτε είχε να κάνει με την ακροτική πολιτική και αυτό το οποίο αναφέρθηκε πραγματικά ε, αναφέρεται σε όλα όσα έχει πει το ελεγκτικό συνέδριο. Πολύ συχνά δεν τα λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή την κριτική της, του ελεγκτικού συνεδρίου για οτιδήποτε έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι τα χρήματα του φορολογουμένου θα πρέπει να αποτελέσουν, ε, ε, να δίνονται με βάση τα έσοδα ε, και τα έξοδα του αγρότη. Θα πρέπει τα δημόσια χρήματα να σχετίζονται με τα αποτελέσματα και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μελλοντικά αναπόσπαστο κομμάτι της ΚΑΠ. Και εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσουμε ακριβώς τα όσα λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Νιέγερτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή, τον κύριο Λαβία. Είναι πολύ καλή η έκθεσή του. Πολύ ισορροπημένη. Και τροφή προς περαιτέρω συζητήσεις στην Επιτροπή Γεωργίας για τις προτάσεις που κάναμε για μεταρρυθμίσεις. Να ξεκινήσω αναφερόμενος στη γενική αρχιτεκτονική. Ποιος είναι ο στόχος μας. Βλέποντας την παρούσα ΚΑΠ, συμπεράναμε ότι μια γενική προσέγγιση για όλη την Ένωση που έχει 28 κράτη-μέλη με πολύ διαφορετικές κλιματολογικές και αγροτοοικονομικές συνθήκες είναι κάτι που δεν λειτουργεί. Αυτή ήταν η βασική μας αξιολόγηση και η πρόταση μεταρρυθμίσεων που υποβάλαμε ξεκίνησε από εκεί. από το νέο μοντέλο βάσει αποτελεσμάτων, όσοι σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας. Θέλουμε να απομακρυνθούμε από την απόλυτη συμμόρφωση, δηλαδή ένα σύστημα βασίζεται αποκλειστικά στη συμμόρφωση, να κάνουμε κάτι που λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις. Δεύτερον, θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη επικουρικότητα στα κράτη-μέλη, να αποφασίζουν τις παρεμβάσεις και τα μέτρα που θέλουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τρίτος πυλώνας. Όλα αυτά θα πρέπει να καταλήγουν σε απλούστευση απλό σύστημα και για τους γεωργούς και τις εθνικές αρχές. Τώρα αυτό που οδηγεί σε 27 εθνικές αγροτικές πολιτικές ή επανεθνικοποίηση. Η άποψή μας είναι στα εναρή. Λέμε όχι. Θέσαμε ένα πλαίσιο. Κυρίσταν παρόδο κάτι που υποστηρίζει και η νομική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Οι πυλώνες αυτοί είναι κοινοί για όλα τα κράτη-μέλη. Κοινή στόχη για πρώτη φορά που θα αναφέρονται ρητά στους κανονισμούς μας. Θα υπάρχει ένα κοινό σύστημα δικτών και υπάρχει ισχυρότατο σύστημα διακυβέρνησης του κανονισμού. Έτσι τα κράτη-μέλη θα καταθέτουν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σαφέστατους στόχους και θα εγκρίνονται αυτοί οι στόχοι μόνο αν ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες και τους στόχους που από κοινού θα έχουμε θέσει. Ένα συγκεκριμένο σημείο πρότεινε ο κύριος Λαβία και δείχνει την προσέγγισή μας. Είπατε ότι θα πρέπει να ε, βάζουμε μια, ένα κατάλογο με οικολογικά συστήματα βάσει κατά εξουσιοδότηση πράξεων. Όταν είδαμε την προσέγγιση για το πρασίνισμα, είδαμε ότι τελικά δεν είμαστε εμεί σοφότεροι στον φάτο πρασίνισμα. Ίσως να είσαι καλύτερη θέση στα κράτη-μέλη να δουν τι θα μπορούσε να είναι αποδοτικό με συγκεκριμένο στόχο και δίνει αποτελέσματα ε, στη δική τους χώρα, στη δική τους ύπεθρο. Δεν πρέπει να περιορίζουμε τα κράτη-μέλη, να του αφήσουμε ευχέρεια κινήσεων. Και γι' αυτό στα οικολογικά συστήματα βάλαμε ένα πλαίσιο υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε στην τρέχουσα περίοδο για το πρασίνισμα. ακριβώς ε, τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και ακριβώς τι πρέπει να κάνουν οι γεωργοί. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον. Τις πυλώνες ακολουθούμε. Για ό,τι σχετίζεται με άμεσες πληρωμές και αυξημένη αρεσιμότητα λέμε ότι όλοι οι γεωργοί θα πρέπει να συμμορφωθούν στην Ευρώπη και αυτό ισχύει και το παρόν σύστημα διασταυρωμένης συμμόρφωσης και κάποια στοιχεία παίρνουμε από το σύστημα πρασινίσματος και έχουμε όμως προβλέψει και την κατάλληλη ευελιξία για τα κράτη-μέλη για να λάβουν υπόψη τις διάφορες ιδιαιτερότητες τους. Δεύτερος πυλώνας, υποχρετικά συστήματα δυνάμει του πυλώνα 1 και 2, τα οικολογικά σχήματα δεν θα είναι θελοντικά, θα είναι για τους γεωργούς αλλά όχι για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα υποχρεούνται να κάνουν κάποιες προσφορές στους ε, γεωργούς πάνω σε αυτό Και τα έχουμε περιβάλει όλα αυτά λέγοντας ότι το άρθρο 92 προβλέπει νομική υποχρέωση για τα κράτη-μέλη στο στρατηγικό πλαίσιο της ΚΑΠ να αποδεικνύουν ότι επιδιώκουν ε, ένα στόχο πολύ φιλόδοξο για την προστασία του περιβάλλοντος και ε, την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Όλα αυτά είναι μια στέρεη βάση για την επίτευξη περισσότερων αποτελεσμάτων για την προστασία του περιβάλλοντο και περισσότερα μέτρα για την μείωση των αποτελεσμάτων αλλαγή αλλαγής του κλίματο. λαμβάνοντα υπόψη και τα μαθήματα που αποκομίσαμε από τα ισχύοντα. Τώρα, μεταφορά μεταξύ πυλώνων. Κατανοώ τη θέση σα. Αυτό σχετίζεται με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Άλλοι φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώση ασχοληθούν με αυτό και θα μα πούν τι θα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να προσέξουμε κάτι όμως το ότι προτείνεται να μην υπάρξουν αλλαγέ από τον ε, πυλώνα 2 προ πυλώνα 1 για μεταφορέ εκεί, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερη προστασία για το περιβάλλον και καλύτερη καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο. Στο πρώτο πυλώνα υπάρχουν τα οικολογικά ε, προγράμματα και πλαίσια. Μπορεί να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη ότι θα εστιαστούν περισσότερο στα συστήματα αυτά και θα πρέπει να θέσουν εκεί περισσότερα χρήματα και τότε θα μπορεί να υπάρξει η αναγκαία ε, ευελιξία για τη μεταφορά μεταξύ πυλώνων. Μετά το άλλο θέμα, εξολόγηση αντικτύπου και τη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όλοι γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει στεναρά τι κατηγορίες του ελεγκτικού συνεδρίου που αναφέρει στη γνωμοδότηση ο Επίτροπος Χόγκαν είπε, το είπε αυτό δημοσία και ήταν της σχετική του παρέμβαση στην Επιτροπή Γεωργίας. Τούτου λεχθέντος έχουμε γραπτό προβεί ανάλυση σημείο προ σημείο και αναλύουμε την γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου και είπαμε ότι πραγματικά υπήρξαν κάποιες παρερμηνίες και παρεξηγήσεις σχετικά με τους στόχους μας. Στείλαμε επιστολή και στο Συμβούλιο και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και με τα χαράς να στείλουμε και σε εσά αντίγραφο για να διατρέξετε το κείμενο και να δείτε τη λεπτομερή απάντηση που δώσαμε στο ελεκτικό συνέδριο. Για την αξιολόγηση αντικτύπου έχουμε μια τέτοια ανάλυση με παρελές εκατοντάδες ε, σελίδες. Μία από αυτές τι αναλύσεις συνοδεύει και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε. Τέλος, για το πότε θα αρχίσει η μεταρρύθμιση. Πιστεύω μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί στους αγρούς και στις εκμεταλλεύσεις το ταχύτερο δυνατό. Ελπίζουμε να έχουμε και εκεί καλύτερες υψηλότερες φιλοδοξίες και να μην καθυστερήσουμε το 2023. Αλλά πολύ προηγουμένως, πολύ πιο νωρίς αυτό να εφαρμοστεί για τους γεωργούς. Ευχαριστώ ο εισηγητής ο κύριος Λαβία λοιπόν να ολοκληρωθεί η συζήτηση από αυτού. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ποικιλία των παρεμβάσεών τους και των απόψεών τους. Όλα αυτά δίνουν σε μένα και σε μας συμπληρωματικά στοιχεία που μπορούν να προσανατολίσουν τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην Επιτροπή. Επιτρέψτε μου να απογραμμίσω μία-δύο πτυχές από αυτές που άκουσα κάποια σημεία που βρίσκουν σύμφωνα, όπως ενίσχυση του χαρακτήρα του περιβαλλοντικού και διασύνδεση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα και της πολιτικής πληρωμών. Και από την άλλη πλευρά, να υπενθυμίσω εν πρώτης και σε μέναν πρώτα απ' όλα κάτι. Και για να το ακούσουν συνάδελφοι, όλη η δουλειά που κάναμε σε αυτή την Επιτροπή για την καταπολέμηση αλλαγή του κλίματος και για την προστασία του περιβάλλοντος σε τομείς διαφορετικούς δεν είναι ε, να τεθούν όρια όσον αφορά την παραγωγή την ενεργειακή και την παραγωγή τη βιομηχανική. Δεν είναι διανοητό να το κάνουμε αυτό χωρίς να συμπεριλάβουμε το γενικό τομέα στην καταπολέμηση ε, της αλλαγής του κλίματος, στον αποτεσμό της αλλαγής του κλίματος και στην προστασία του περιβάλλοντος και η δική μας πολιτική, η γεωργική πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να συμβάλλει στη γενική προσπάθεια. Πώς υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Εγώ εξέφρασα μια άποψη. Βλέπω ότι κάποιοι συνάδελφοι τίνουν να πιστεύουν ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν καλύτερο να, καλύτερα να προσαρμοστούν με επιλογές που θα γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Και αυτή είναι προφανώς και η άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ πιστεύω ότι η πρόταση το να δημιουργήσει μια, ένα ευρύ πλαίσιο μέσω κατά εξισοδότηση πράξεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιες επιλογές να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορεί τα κάτι μελη να επιλέξουν, αλλά θα υπάρχει μια ομάδα προτάσεων που θα έχουν αποτελέσματα και από εκεί θα επιλέγουν τα κάτι μελη Εγώ Πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα η προστασία του περιβάλλοντο και την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Γι' αυτό έκανα αυτή την πρόταση. Ε, από όλου του συναδέλφου ακούστηκαν ενδιαφέρουσε προτάσει, θα τι αξιολογήσουμε. Και καταλαβαίνω αυτό που προσπαθούν να πούν. Και πού συμφωνούν με τον εισηγητή. Ελπίζω όμως να μην λάβω τεράστιο αριθμό τροπολογιών μετά από όλα αυτά που θα περιπλέξει τις εργασίες μας. Και μετά θα μας δυσχεράνει από πλευράς χρονικής. Συμφωνήσαμε και με τη Γραμματεία Πρόεδρε να θέσουμε προθεσμία για τις τροπολογίες. 11 Δεκεμβρίου θα είναι η προθεσμία. 11 Δεκεμβρίου. Επιτρέψτε μου να ζητήσω, αφού συνομιλήσω με όλες τις πολιτικές ομάδες και υπό το φως του ότι κατανοώ ότι υπάρχει μια συγκέντρωση πολλών εκθέσεων, διότι όλοι πάμε στην Ολομέλεια του Απριλίου, με πάρα πολλές εκθέσεις την ίδια περίοδο. Και οι πιο πολιτικές ομάδες, οι μικρές πολιτικές ομάδες, που έχουν και πιο ε, μικρό αριθμό προσωπικού, έχουν μεγάλες δυσκολίες. Ζητώ μερικές ημέρες παραπάνω και να πάμε στην παλιά ιδέα 13 του μηνό να, κάνουμε, να βάλουμε την προθεσμία στις τροπολογίες. Έτσι να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη όλες τις προτάσεις και πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμες και θα, θα συμβάλλουν στην προσπάθεια και στο τέλος θα έχουμε μια ισχυρή γνωμοδότηση της Επιτροπής μας να την υποβάλουμε στην Επιτροπή Γεωργίας μετά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαβία. Όντως, 13 Δεκεμβρίου έχουμε μια παράταση της προθεσμίας ελπίζοντας να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ε, τέλη Φεβρουαρίου. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής και την Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη το 2019. Έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του κύριου Κόβατσεφ, στον οποίο δίνω και το λόγο. Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός και να σας εξηγήσω τα βασικά στοιχεία του σχεδίου γνωμοδότης. Όπως ξέρετε, η Τήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη ε, εγκαινιάζει το νέο ε, κύκλο οικονομικής, ε, οικονομικού συντονισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξαμήνου και πέραν της οικονομικής πολιτικής παρακολουθούμε και τους, τις πολιτικές μας υπό τη σκοπιά των στόχων το, της βιώσιμης και είναι σημαντικό η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να προσαρμόζεται σε ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμη στρατηγική ε, που θα καθοδηγείται από του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. και θέλουμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη προκειμένου να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μάλλον ε, ε, περιβαλλοντικά βιώσιμο και, περιβαλλοντικά βιώσιμο και κοινωνική ανάπτυξη χωρί αποκλεισμού. Επίση, θέλουμε βιώσιμε προποθέσει για ανάπτυξη και επενδύσει στον τομέα αυτό. Ε, γενικώ είμαστε υπέρ τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί σε βασικέ προτεραιότητε, αλλά μην ξεχνάτε ότι η οικολογικοποίηση τη οικονομία και η επένδυση σε πιο αποτελεσματικά συστήματα υγεία θα αυξήσει και την ανταγωνιστικότητά μα ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύσει και θα ενισχύσει την υγεία και την ευημερία των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι σημαντικός μηχανισμός για την προώθηση των βασικών και απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και από την άποψη αυτή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σαφή σύνδεσμο μεταξύ τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού και των συστάσεων για τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που εντοπίζονται στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ο σύνδεσμο όμω αυτό, η διασύνδεση αυτή, θα πρέπει να λάβει τη μορφή τη αιρεσιμότητα, γιατί μερικέ φορέ χρειάζονται χρόνια για να φανούν τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων. Οπότε χρειαζόμαστε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική σε αυτή την αξιολόγηση. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη τι στάσει μα από προηγούμενε χρονιέ στα πλαίσια τη υγεία, των υπηρεσιών υγεία και σίγουρα περάσαμε από ε, τις οικονομίες σε μια ε, προσέγγιση που εστιάζεται περισσότερο στις επιδόσεις των συστημάτων υγείας. Θα πρέπει να γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε τη σημασία της υγείας και την ανάγκη για ποιοτική υγεία. Δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στα οικονομικά στοιχεία, γιατί κάτι τέτοιο θα υποσκάψει την βιωσιμότητα. Επίσης, αν δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε την ε, το φιλόδοξο πρόγραμμά μας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη χωρίς υγιείς συμπολίτε χωρί υγιεί Ευρωπαίου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επικεντρωνόμαστε και στι επιδόσει των συστημάτων υγεία. Ευχαριστώ και περιμένω ε, τι προτάσει των ε, σχεδόν εισηγητών. Εκ μέρου ε, του σχεδόν εισηγητού ε, του κυρίου Σορίνιο. Θα μιλήσω εγώ, ζητώ συγγνώμη από το σκιώδη συγητή, από, εκ μέρους του σκιώδη εισηγητού που μου ζήτησε να παρουσιάσω τι παρατηρήσει του. Καταρχήν, να τον κύριο Κόβατσεφ για το σχέδιο γνωμοδότηση. Ο κύριο Ζωρίνιο σε μεγάλο βαθμό συμφωνεί με τον εισηγητή, παρόλο που θα καταθέσει και επιμέρου τροπολογίε. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να υπογραμμίσουμε περαιτέρω την κλιματική και περιβαλλοντική πολιτική που θα πρέπει να διαδραματίζει ε, ένα ρόλο που θα λαμβάνει υπόψη και τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επίση, να συμπεριληφθεί ο στόχος της ε, μιας οικονομίας που θα είναι ουδέτερη για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επίσης, να διατρανώσουμε την δέσμευσή μας ε, για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 μέσω μιας δίκαιης μετάβασης, κοινωνικά δίκαιης ε, και αποτελεσματικής απόψη κόστους. Επίσης, με τις τροπολογίες ο κύριος Ζωρίνιο θα προτάξει την ιδέα της δίκης μετάβασης που θα προσαρμόσει τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού προκειμένου να μειώσουμε τον αντίκτυπο που θα έχει στην απασχόληση η απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Επίσης, ζητούμε συμμετοχή, συγκροτημένη συμμετοχή των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Αξιάμινο και μεγαλύτερη συμμετοχή και των Υπουργών Περιβάλλοντος στην διαδικασία αυτή σε επίπεδο Συμβούλιου. Σας ευχαριστώ. Αυτά από τον κύριο Ζωγίνιο, τον Σκιώδη Συγητή. Ευχαριστώ κύριο Εκχότ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ πολύ λακωνικό. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κόβατσεφ, για το σχέδιο γνωμοδότησή του. Πιστεύω ότι περιέχει πολλά καλά σημεία και θετικά που μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Ε, θα το ενισχύσουμε, θα ενισχύσουμε την γνωμοδότηση αυτή, θα τη συνδέσουμε με τα εθνικά ε, σχέδια για την ενέργεια ε, να το συνδέσουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό το χαρακτήρα θα έχουν οι τροπολογίε μα. Συμφωνώ να το συνδέσουμε με τον κοινωνικό πυλώνα, με το στόχο βιώσιμη ανάπτυξη, όπω προτείνετε κι εσεί. Μόνο το θέμα τη αιρεσιμότητα δεν μα βρίσκει σύμφωνο. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον τρόπο που το διατυπώνετε. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μορφή αιρεσιμότητα. Θα δούμε πώ θα το διατυπώσουμε με έξυπνο τρόπο και πώ θα το εφαρμόσουμε με έξυπνο τρόπο, ώστε να μην πλήξουμε φυσικά τον κόσμο αλλά η συζήτηση περί ερεσιμότητας θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Και από αυτή την άποψη η γνωμοδότηση σας χρήζει κάποιες μικρής ε, Κατά το λοιπόν όμως συμφωνούμε. Ευχαριστώ κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν... Ε, βλέποντας την έκθεση της Επιτροπής, διαπιστώνω με μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα και στην Γαλλία, ότι τονίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης της φορολογικής δικαιοσύνης και μάλιστα διάβασα μία παράγραφο που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Τη στιγμή της παγκοσμιοποίησης, την, εποχή της παγκοσμιοποίησης, η ικανότητα της ε, μιας κυβέρνησης να επιβάλλει ε, τους μεγαλύτερους ε, μισθούς είναι περιορισμένη. Θέλουμε μία ε, δίκαιη φορολογία, λαμβάνοντας υπόψη και την ψηφιακή οικονομία. Αυτό είναι προϋπόθεση για να έχουμε ε, μία ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Και βλέπετε τι γίνεται από τα γεγονότα στη χώρα μου, γιατί οι πολίτες θέλουν να καρπώνονται περισσότερο τα πλεονεκτήματα και της ε, ψηφιακής οικονομίας. Ήταν λάθος λοιπόν να γνωρίσουμε αυτό το στοιχείο και πραγματικά δεν θα το καταλάβουν οι πολίτες, ιδιαίτερα στην προεκλογική εκστρατεία. Θέλουμε ένα πλαίσιο που θα είναι πρόσφορο για τις ε, βιώσιμες, ε, για τις λαμβάνοντας υπόψη όμως την ανάγκη βιωσιμότητας. Επίσης έρευνα, καινοτομία, τεχνολογική ανάπτυξη, ψηφιακές τεχνολογίες τι γίνεται όμω με τη βιομηχανία, δεν μου λέτε τίποτα. Θα εγκαταλείψουμε το δευτερογενή τομέα. Καταλάβαμε ότι η ψηφιακή, τεχνολογική και ενεργειακή μετάβαση ε, δεν είναι άειλη. Χρειάζεται μεταποιημένες πρώτες ύλε. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποποιηθούμε τελείως ε, την ανάγκη της επαναβιομηχανοποίησης της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς παρακαλώ. Όχι. Οπότε επανερχόμαστε στον κύριο Κόβατσεφ. Όχι, συγγνώμη, προηγουμένω να ακούσουμε την κυρία Βέκη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και του συναδέλφου που ζήτησαν το λόγο. Εντάχει, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία και ευχαριστώ για τα σχόλιά σας σχετικά ε, με την ε, ετήσια έρευνα και την ανάπτυξη θα τα λάβουμε υπόψη μας ε, όλα αυτά και ότι θα μεταβιβαστούν αυτά και στο Συμβούλιο όπου θα συζητήσουν το θέμα αυτό, την έρευνα αυτή ε, του χρόνου. Χαιρόμαστε ε, για το γεγονός κάποια θέματα όσον αφορά την υγεία, την βιωσιμότητα περνούν ε, και ότι ε, έχουν ε, πιο κεντρική θέση για την φετινή έρευνα. Βρισκόμαστε σε καλή θέση, θα πρέπει να, να το θυμόμαστε αυτό. Έχουμε την έκτη χρονιά κατά, στη σειρά με ανάπτυξη. Έχουμε μειωμένη ανεργία μεταξύ των νέων. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό. Αυτό βέβαια όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε εξοπλισμένοι για τις μακροπρόθεσμες ε, προκλήσεις οι οποίες εμφανίζονται και γι' αυτό το λόγο έχει έρθει η ώρα να δράσουμε ε, και φυσικά η συμπερίληψη και η βιωσιμότητα είναι δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία τονίζουμε στην έρευνά μας και όσον αφορά τα όσα είπε η κυρία Γκροστέτ ε, και ο εξυγχρονισμός ε, των βιομηχανιών μας αναφέρεται διότι θεωρούμε ότι και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο ε, της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία και της μείωσης των εκπομπών και το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους συναδέλφους αλλά και την Επιτροπή για τα σχόλιά τους. Συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα υπόθηκαν ε, την πολιτική για το περιβάλλον, για τις κλιματικές αλλαγές. Ε, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με την τεχνολογική επανάσταση, με την... θα πρέπει να έχουμε καινοτομία, όθηση της οικονομίας, να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών, ε, μέχρι το 2050 να φτάσουμε τις μηδενικές εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα όσον αφορά την ερωσιμότητα δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν οι πολίτες μας και οι περιφέρειές μας. Θα πρέπει να βρούμε έναν ε, τρόπο ώστε να υπάρξει αυτός ο σύνδεσμος. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και θα χαρώ να συζητήσουμε περαιτέρω την συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Η Προθεσμία είναι η 9η Ιανουαρίου ε, μέχρι τις 11 η ώρα ε, για την υποβολή ε, τροπολογιών θα πρέπει να είναι στα αγγλικά. Και στις 25-26 θα Φεβρουαρίου θα ακολουθήσει η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Και περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, της συζήτηση σχετικά με την απαλλαγή του Γενικού Προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την Ευρωπαϊκή Αρχή, για την Ασφάλεια Τροφίμων, Οργανισμό Περιβάλλοντος, Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, Οργανισμό Φαρμάκων, Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Θα ξεκινήσω λοιπόν κάνοντας κάποια σχόλια. Όπως και τα προηγούμενα έτη, η ΕΝΒ θα καταθέσει συνολικά έξι νομοδοτήσεις. Όσον αφορά τώρα την Επιτροπή, φέτος το ε, ελεγκτικό συνέδριο δεν παρήχε ένα συνολικό ε, ποσοστό λάθους ε, σχετικά με την αλληλεία, την κλιματική δράση. Ανταυτού όμως μας παρουσίασε τα λάθη τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν σε αυτόν τον τομέα όπως για παράδειγμα μη επιλέξιμη δικαιούχη, ε, δράσεις, ε, δαπάνες. Όσον αφορά συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον το 2017, το LIFE, ε, το πρόγραμμα αυτό, γιόρτασε τα 25 χρόνια, έδωσε 225 ε, ε, ευρώ για να ε, χρηματοδοτήσει 100 νέα προγράμματα. Όμως θα πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες ούτως ώστε να μειωθούν οι επενδύσεις και σε αυτό το πλαίσιο το 5 με 8% των πληροπών ξεπέρασαν τις προθεσμίες για το 2017 σε σχέση με ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 3,9% για το 2019. Επίσης, η μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του LIFE έγινε το 2017, όμως κατά τη διάρκεια της περίοδου που καλύπτονταν ε, για την αξιολόγηση 14 με 15, πολλά προγράμματα ακόμα έπρεπε να ξεκινήσουν ενώ ελάχιστα είχαν ολοκληρωθεί όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον. Οι βασικότερες ανησυχίες ε, αφορούν τον ε, στόχο 20% για την προστασία του κλίματος ε, στο πλαίσιο του ΠΔΠ και δεν καλύφθηκαν για το 2017 καθότι μόνο το 19,3% του κοινωτικού προϋπολογισμού ε, καλύφθηκε. Επίσης, όσον αφορά το γεγονός ότι η έκθεση ετήσιας δραστηριότητας ε, της Γενικής Διεύθυνσης του 2017 περιλαμβάνει ε, και αδυναμίες όσον αφορά την ασφάλεια που έχουν ταυτοποιηθεί στο πρόγραμμα ανταλλαγής εκπομπών. Όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, ολοκλήρωσε μια ενδιάμεση αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος υγείου, το οποίο συμπεριέλαβε, τόνισε μάλλον την ε, σχέση για ε, των αναγκών των κρατών ε, μελών και πρότεινε την ενίσχυση των ε, προσπαθειών της ε, Ένωσης. Επίσης, ε, τονίζει το μέσο ποσοστό λάθους στο 2,5% το οποίο είναι πάνω από το όριο του 2%. Γνωρίζουμε ότι αυτό αφορά τις υπερδηλώσεις της αιτήσει πληρωμών λόγω διαρθρωτικών αλλαγών που έγιναν στην διαχείριση και τους ελέγχους των των αιτήσεων από ένα κράτος ε, μέλος. Ε, ζητούμε λοιπόν από την ε, Γενική Διεύθυνση να μην επαναληφθεί αυτό μελλοντικά. Όσον αφορά τώρα τις υπηρεσίες, οι εκθέσεις εξετάζουν το πώς έχουν χρησιμοποιηθεί οι πόροι, τόσο όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς πόρους, αλλά και το προσωπικό σε αυτό το πλαίσιο. Ένα γενικό σχόλιο είναι ότι με κάποια, κάποιες αποδόσεις δεν μπόρεσαν να παραδοθούν το 2017 για κάποιες υπηρεσίες λόγω των των ε, περιορισμών στους ε, πόρους. Οι γνωμοδοτήσεις επίσης τονίζουν τα, ε, βασι, τις βασικές ε, επιστημονικές και τεχνικές αποδόσεις και το σημαντικό είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο ξεκίνησε, δήλωσε μάλλον, ότι οι ετήσιοι ε, λογαριασμοί για το 2017 είναι όλοι ε, νόμιμοι και τακτικοί και με βάση τα δεδομένα αυτά ε, θα, θα συστήνεται μάλλον ότι θα υπάρξει εκφράζεται ικανοποίηση σχετικά με την, με την εφαρμογή του προϋπολογισμού από την Επιτροπή και οι εκθέσεις εκφράζουν λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, παρασχεθεί απαλλαγή ε, στην Επιτροπή και στις ε, πέντε υπηρεσίες υπό την εντολή της ΕΝΒΗ και τώρα θα χαρώ να ακούσω από τους συναδέλφους, από τους Κεώδης η κυρία Κάντενμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Βάλεαν ε, για το έργο της ε, και για τις έξι γνωμοδοτήσεις που αφορούν την απαλλαγή του 2017 για διάφορες υπηρεσίες για τις οποίες είναι συνυπεύθυνη και η Επιτροπή ΕΝΒΗ, ΕΦΣΑ, η ΕΜΑ, EA και ΕΧΑ και στο πλαίσιο της ε, Επιτροπής Μπάτς ε, ως σκιώδης ε, είμαι υπεύθυνη για κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες οπότε είναι θέματα τα οποία γνωρίζω καλά. Συνολικά λοιπόν και ο γενικός προϋπολογισμός για την DG Sante κλίμα καθώς επίσης και για τις πέντε υπηρεσίες θα πρέπει να δοθεί απαλλαγή. Δύο σχόλια επιπλέον. Το πρώτο όσον αφορά τη γνωμοδότηση για τον γενικό προϋπολογισμό να προσθεθεί μία ακόμα παράγραφος όσον αφορά ε, την εφαρμογή του προγράμματος για την προστασία των φυτών και της ε, εργασιακής ε, υγείας και ότι εφαρμόστηκαν όλες οι πληρωμές ορθά και επίσης να προσθέσουμε μία παράγραφο ότι πολλά από τα μέτρα του προγράμματος υγείας ε, στο πλαίσιο της υπηρεσίας ε, για, τα, ε, για την προστασία των τροβίμων εφαρμόστηκε πλήρως. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο όσον αφορά το πώς θα διατυπωθεί και το πώς θα συμπεριληφθεί, αλλά θα ήθελα να γίνει στην παράγραφο 14 τώρα σχετικά με τις ε, σχετικά με το ποσοστό λάθος της Γενικής Διεύθυνσης ε, σάντε, θα ήθελα να πω ότι αυτό ε, τονίστηκε από τα κράτη-μέλη και επεξεργάζεται περαιτέρω. Τώρα όσον αφορά την ΕΚΑ θα ήθελα να αναφέρω ότι και εδώ έχουμε διάφορες εταιρείε οι οποίες κατά λάθος οι επειδή δεν ξέρουμε κάναν κάποιες λάθος δηλώσεις οπότε θα πρέπει εδώ να γίνει, έγινε περαιτέρω έλεγχος με αποτέλεσμα να έπρεπε να γίνει γίνουν περαιτέρω έλεγχοι, το οποίο αύξησε το κόστο. Όσον αφορά την ΕΦΣΑ θα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο και αν συμφωνεί την πρόταση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, τότε θα έχουμε αυξημένα ε, κόστη ε, για την ΕΦΣΑ. Γνωρίζω ότι από τη μία πλευρά πρόκειται για ε, μία έκθεση απαλλαγής, παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι για το έργο της ΕΦΣΑ θα χρειαστούν περαιτέρω κονδύλια, ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκροστέτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα όλα όσα μας παρουσιάσατε. Θέλω να τονίσω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Η απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ελπίζω ότι οι τροπολογίες που ίσω κατατεθούν θα πρέπει παραμένουν επί θεμάτων δημοσιονομικών και να μην είναι πρόσχημα ούτω ώστε μέσω τη απαλλαγή να παρέμβουν στι εργασίε του οργανισμού. Να επιστήσω την προσοχή όλων των συναδέλφων επί του σημείου 4 τη νομοδοτήσεω σα, κυρία, κυρία Βαλιάν, την οποία υποστηρίζω πλήρω και υπογραμμίζει το θέμα των πόρων του οργανισμού. Και έχετε δίκιο, διότι από τη μια πλευρά του δίνουμε πολλέ νέε αποστολέ, μεταξύ άλλων, και είναι θέμα που ξέρω καλά, ο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα, και από την άλλη πλευρά πρέπει να αντιμετωπίσει ένα κόστο, το κόστο μετακόμιση και την απώλεια προσωπικού για να διαχειριστεί τις πολλές αυτές αλλαγέ μεταξύ των οποίων είναι και σημαντικέ αποστολέ για τη δημόσια υγεία και γι' αυτό είναι επιτακτικό να έχει υπηρεσία φαρμάκων του αναγκαίου πόρου. Και αυτό δεν ισχύει τώρα. Ε, είναι ανεπαρκή η πόρη. Σα υποστηρίζω και πιστεύω ότι είναι σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει γνώση αυτών των δυσκολιών, τι λάβει υπόψη και να αυξήσει τους πόρους του οργανισμού, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ε, στο ύψος των περιστάσεων, δηλαδή να μπορεί να προσαρμοστεί στους νέους στόχους που ανατίθεται. Ευχαριστώ πολύ και του δύο για την υποστήριξή σας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Προσβλέπω λοιπόν στις τροπολογίες σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ήθελε να παρέμβει. Η κυρία Βακρού. Ίσως όμως και κάποιος άλλος εκπρόσωπος να θέλει να μιλήσει. Η κυρία Βακρού ξεκινάει λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Η Γενική Επιτροπή Περιβάλλοντος θέλει να πει ότι μας ικανοποιεί η έκθεσή σας κάναμε μια προσπάθεια να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα live στο βαθμό του δυνατού. Θέσαμε προτεραιότητες ε, την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δηλαδή ουσιαστικά τα προγράμματα κληρονομιάς όπως τα αποκαλούμε της προηγούμενης περίοδου και έτσι να έχουμε αποτελέσματα και στοιχεία με τα οποία θα τροφοδοτήσουμε τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση και τη νέα πρόταση για το live που παρουσιάσαμε φέτος. Στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου υποβάλαν προτάσεις προς έγκριση. Σημειώνουμε αυτά που είπατε για τις καθυστερήσεις των πληρωμών, αλλά έχουμε κάποια δικαιολογία εκεί. Προσπαθούμε να εκτελέσουμε τις πληρωμές με ακρίβεια αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όπως γνωρίζετε ίσως, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό σφάλματος ε, που παρουσιάζεται και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Λαμβάνουμε υπόψη το σχόλιο σας και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε έτσι περαιτέρω. Έχουν γίνει και σημαντικές περικοπές προσωπικού. Πρέπει να το λάβετε και αυτό υπόψη. Το 2018 ήδη λαμβάνουμε υπόψη αυτό που είπατε σχετικά με αυτό. Θα, θα το έχουμε στη Γενική Διεύθυνση, ε, στην έκθεση της Γενικής ως Περιβάλλοντος, στην ετήσια έκθεση αυτό. Προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία και συντονισμό για να παρουσιάσουμε ε, το πρόγραμμα LIFE ε, που θα έχει πετύχει καλά αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Νίκ Φωνόρμακ από το τμήμα υπεύθυνο για τις δράσεις της Γενικής Δευθύνσεως Περιβάλλοντος. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν γνωμοδότηση. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό, για τα θέματα που αναφέρθηκαν, για να ληφθεί υπόψη η διάσταση του κλίματος σε όλες τις πολιτικές. Δεν φτάσαμε ακόμα στο στόχο. Υπάρχουν πιθανότητες μέχρι το 2020 να πετύχουμε αυτό το πολύ φιλόδοξο στόχο. Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια από όλου του ενδιαφερομένου, όλους του εφαρμοστικού φορείς για να πετύχουμε το στόχο. Σωστός ο δρόμος που ακολουθούμε. Είμαστε πρωτοπόροι. Το σχέδιο προπολογισμού του 2019, που σύντομα θα είναι τελικός προπολογισμό για το 2019, λαμβάνει υπόψη τη συμπερίληψη του κλίματος και έχει αυξηθεί το κονδύλι κατά 20,1% ε, και πρέπει να καταρτιστεί και ο προπολογισμό του 2020. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα και ο κίνδυνος βέβαια αν θα πετύχουμε τον τεθέντα στόχο ή όχι. Για το σύστημα εμπορίου ρήπων, το ETS τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, είναι ένα σύστημα με κίνδυνο. Είναι κάτι σαν σύστημα του τραπεζικού τομέα και γι' αυτό θέλουμε και πρότυπα κατάλληλα να υπάρχουν και τα συγκρίνουμε και τα πρότυπα που θέλουμε να θέσουμε εδώ με αυτά του τραπεζικού τομέα. Έχουμε υλοποιήσει κάποιε δράσει σε ένα σχέδιο δράση, πολύ διευρυμένο. Μετακινήσαμε το σύστημα σε πιο ασφαλείς servers στο Λουξεμβούργο και κάνουμε και κάποια αξιολόγηση κινδύνου. Θέλουμε να δούμε ποιο κίνδυνο, απομένει, ποιο επίπεδο κινδύνου απομένει μετά την εφαρμογή του σχεδίου δράση. και από αυτό εξαρτάται αν θα άρουμε την επιφύλαξή μα από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2018. Αυτό είναι ένα από του όρου για την άρση της επιφύλαξης. Δεν μπορώ όμω να προδικάσω ποια θα είναι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Ευχαριστώ. Άλλος. Εγώ θα είμαι τελευταίο. Από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας. Η δική μας Γενική Διεύθυνση χαιρετίζει φυσικά το σχέδιο γνωμοδότησης που είναι σαφέστατο. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα για την ασφάλεια τροφίμων και την υγεία, έχουμε σχεδόν πλήρη εκταμείευση και τηρήσει τη ανάληψη υποχρεώσεων για το 2017. Για το ποσοστό σφάλματος, αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα το νέο δημοσιονομικό κανονισμό που προβλέπει δυνατότητα απλούστευση στην επιστροφή του κόστους που έχει αναλυφθεί από τα κράτη-μέλη, ε, ώστε να είναι πιο εύκολα και απλά τα πράγματα και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να γνωρίζουμε τα ποσά που θα επιστρέφουμε για το κόστος που έχουν πραγματοποιήσει, τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει τα κράτη-μέλη. Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφή, ε, Φαρμάκο, συγγνώμη, ε, σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα το 2018-2019. Είναι ιδιαίτερε οι αυτές λόγω της μετεγκατάστασης. Έχουμε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με την ελάχιστη των προτεραιοτήτων που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ. Από τους οργανισμούς έχουμε κάποιον εκπρόσωπο. Ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, από τη Γενική, συγγνώμη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, σίγουρα χρειαζόμαστε κατάλληλους πόρους για να ανταπεξέλθουμε στο, στις μεγάλες προκλήσεις και την αύξηση των καθηκόντων μας ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Μάλιστα. Δεν βλέπω άλλο κανένα. Η κυρία Βακρού, μήπως. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την αξιολόγησή της για φέτος. Οπότε στην επόμενη σας έκθεση θα έχετε και το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Οπότε θα έχετε ένα επιπλέον στοιχείο να σχολιάσετε. Πέραν τούτου, συμφωνούμε πλήρως και στηρίζουμε την έκθεσή σας για την απαλλαγή του ε, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και όσο ό,τι αφορά τον Οργανισμό Χημικών, ε, τον οργανισμό χημικών Προϊόντων και τον ε, Οργανισμό Ασφάλεια Τροφίμων σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανονισμών. Μην ξεχνάτε τη διορία για την κατάθεση τροπολογιών που λήγει στις 11 Δεκεμβρίου 5 το απόγευμα. ελπίζοντα ότι θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στη συνεδρίαση τη 21ης και 22ης Ιανουαρίου. Αυτά και καλή σας υπόλοιπη ημέρα και καλή σα όρεξη. Γεια σας.